Μάλλον όχι, να σας πω ότι θα κάνω μια ανακοίνωση με σύσταση η οποία ε, έγινε, έχει υποβληθεί από την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Έχουν παρέλθει 24 ώρες, δεν έχουν προκύψει ε, αντιρρήσεις ε, και βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 105 το κείμενο εγκρίνεται ε, και θα, ε, και θα, θα δημοσιευθεί αύριο 5η 18 Ιανουαρίου του 2018.